Καλημέρα σας. Περιμένουμε γιατί έλειπαν κάποιες κάρτες ψηφοφορίας. Καλημέρα σε όλους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ψηφοφορία. Ξεκινάμε από την ε, γνωμοδότηση της κυρίας Αντινόλφη. Δεν ξέρω αν είστε όλοι έτοιμοι να ψηφίσουμε. Λοιπόν, συμβαστική τροπολογία 1 της συντάκτριας υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 στην επόμενη σελίδα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 στην επόμενη σελίδα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμ... Τροπολογία 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ, κατά, υπέρ και πάλι, κατά, αποχές, επαλήθευση να κάνουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 8. Μισό λεπτό, γιατί δεν δουλεύει η κάρτα μου. Εγκρίνεται το ή άλλως, αλλά θα ήθελα να ψηφίσω. Και δεν μπορώ. Τι συμβαίνει. Λοιπόν, 14 υπέρ, 8 κατά εγκρίνεται. Μπορείτε να ελέγξετε λίγο την κάρτα μου. Τι συμβαίνει. Yeah. Ah. Thank uh, Λοιπόν, 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 61 μαραγκάλ, λέει ο μιλήτρια. 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 52 περιλαμβάνεται στη συμβαστική τροπολογία 10. Γιατί κάποιος με ρώτησε πια και είπα να ψηφίσουμε την 61. 61 εντάξει, 65. Ζουλό, υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για την 65. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Συμβαστική τροπολογία 11. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 82. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 58. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1. Δεν ξέρω αν δέχεσαι την προπολογία υπέρ. Σας παρακαλώ σκόστε τα χέρια σας υπέρ, κατά, αποχές. Να το επαληθεύσουμε για Α, είστε κατά της ε, παρουσίας τη Ποιοι είναι κατά τη παρουσίαση τροπολογίας. Πάνω από δύο, επομένω δεν ψηφίζουμε. Πάμε απευθεία στην 83 λοιπόν. Κατά τμήματα ζήτησαν οι σοσιαλιστές. Πρώτο τμήμα, πρώτο τμήμα της 83 λοιπόν, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται μάλλον, αλλά να το επαληθεύσουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Όχι, πάμε στην τροπολογία 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Υπέρ. Ναι, θέλετε επαλήθευση της προηγούμενης, της 63, άρχεται η ψηφοφορία για την 63, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2, της κυρίας Ward. Είστε υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Ναι. Κατά κάποιος. Ποιοι είναι κατά της προφορικής τροπολογίας. Ένας, εντάξει. Επομένως μπορούμε να την ψηφίσουμε. Προφορική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 76 στην επόμενη σελίδα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα να ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης συνολικά υπέρ, κατά, αποχές, α, συγγνώμη, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, υπέρ, ή μάλλον συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία, η ψηφοφορια περες της ψηφοφορία. 24 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν για τη συνάδελφα την Όλφη. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ψήφισαν και συμμετείχαν στις σκιώδεις ε, συνεδριάσεις. Να πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστώ με τη γραμματεία και ζητώ συγγνώμη από τις πολιτικές ομάδες. Ε, για παράδειγμα με το ΕΛΚΑΝ υπήρξαν παρανοήσεις, αλλά εγώ ποτέ δεν θέλησα να δώσω πολιτικές κατευθύνσει και πριν ειδοποιήσω και υπάρχει συμφωνία με όλους. Νομίζω ότι θα το συζητήσουμε εις βάθος αργότερα στη συνεδρία των συντονιστών και λυπάμαι επίσης που δεν ε, συμπεριλήφθησαν όλοι οι βουλευτές γιατί εμείς είμαστε Επιτροπή του Πολιτισμού. Επομένως πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε τους πάντες ε, στη διάρκεια των συνεδριάσεων των σκιωδών συγητών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω βεβαίως και τη συντάκτρια και του χειώδεις συντάκτες και τη γραμματεία. Ήταν περίπλοκη δουλειά, αλλά νομίζω ότι τελικά καταφέραμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε στην ε, δεύτερη ψηφοφορία. Γνωμοδότηση του κυρίου Χουντή. Δεν ξέρω αν θέλετε κύριο Χουντή το λόγο. Θα μιλήσετε στο τέλο. Ε, εντάξει. Ξεκινάμε. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Συγγνώμη, θέλετε να ψηφίσουμε τη συμβαστική άρχια τη ψηφοφορία. Έλεγχος, λοιπόν, για την ε, συμβαστική τροπολογία 1. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Κομοντίνη, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασ... 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13. Ομπερμάιρ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ, Κατά. Επαλήθευση. Τη συμβιβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Άρα 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Της 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και πάλι. Ισοψηφία. Α, κάνετε λάθος, αλλά ούτως ή άλλως δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Ή μάλλον δεν είναι το ίδιο. Έχει κλείσει όμως ψηφοφορία, λυπάμαι. 16 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 κατά τμήματα κατόπιν αιτήματος του ΕΛΚ. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Θέλω να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται μάλλον. Ναι. Και πάλι με ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 του εισηγητή ε, κατά τμήματα κατόπιν εκείνων των σοσιαλιστών. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και πάλι, λόγω ισοψηφίας. 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33, Ντράγκητσι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές Εγκρίνεται μάλλον, αλλά πρέπει να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 4. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. 36. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές. Να το επαληθεύσουμε. Δεύτερο τμήμα της 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν σε 35. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 39, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 24, Η 40 καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε η 36, δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. 35 την τελειώσαμε, 39 τελείωσε 24. 24. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 42 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται μάλλον, αλλά να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 42. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη 48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 στην επόμενη σελίδα με προφορική τροπολογία του ΕΛΚ. Δέχεστε την προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε η ψηφοφορία. «26 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και μία αποχή μία αποχή. Συγχαρητήρια στο συντάκτη και στους σκιώδεις φυσικά. Δεν ξέρω αν ο συντάκτης γνωμοδότησης θέλει να πει δύο λόγια. Παρακαλώ κύριε Χουντή. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που όχι μόνο που ψήφισαν, υπερψήφισαν την γνωμοδότηση, αλλά γιατί στη φάση των συμβιβαστικών τροπολογιών ε, επέδειξαν, επέδειξαν και όπως και εγώ προσπάθησα να βρούμε ένα κλίμα συνενετικό ούτως ώστε το κείμενο να μας εκφράζει όλους. Ε, με αυτή την έννοια ευχαριστώ πολύ και τους βοηθούς μου την κυρία Λεοτσάκου και τον κύριο Σαμπανόπουλο διότι κατέβαλαν και αυτή προσπάθεια όπως και το επιτελείο μας γιατί καμιά φορά οι αφανείς είναι πίσω από εμά που έχουν κάνει ουσιαστική δουλειά. Εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν δύσκολο κείμενο, θέλω να πω, το είδατε σε κάποιες ψηφοφορίε. Αφού τα καταφέραμε όλοι μαζί στο τέλος, ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να έχει επιτυχία και η εφαρμογή αυτού που εμείς προτείνουμε και γνωμοδοτούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, σας ευχαριστώ γιατί ε, κατάλαβα ότι έγινε τεράστια προσπάθεια από όλου προκειμένου να βρεθεί συμβιβασμός και ευχαριστώ πολύ λοιπόν και για τη δεσμευσή σας και για τους ε, σκιώδη συντάκτες και να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για την συνδρομή της βεβαίως και όλους τους συνεργάτες σας. Ωραία. Τώρα περνάμε στην έκθεση... Μισό λεπτό, συγγνώμη. Για ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ε, μια πολύ μεγάλη μάχη που δόθηκε ε, προκειμένου το 2018 να ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που έδωσαν μάχη για να ε, ε, έχουμε το 2018 σε 18 έτος. Ε, ξέρουμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβλήθηκε πολύ καθυστερημένα, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, με τους συντονιστές και την, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και την Επιτροπή συγγνώμη, αποφασίσαμε να έχουμε μια πιο ταχεία διαδικασία, λίγο πιο απλουστευμένη. Κάποια στοιχεία λοιπόν θα προχωρήσουν λίγο πιο γρήγορα. Εμείς ε, γνωρίζετε λίγο και τη διαδικασία, ε, πρέπει να προχωρήσουμε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, τον κύριο Διακόνου, ο οποίος ήδη ήρθε σε επαφή με τους κοιόδη συζητητές. Ε, θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε για να μπορέσουν όλοι να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η προστασία και η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ε, θα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί και οι πολιτιστικές προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο. Ε, ξέρουμε ότι υπήρξαν κάποιες καινοτομίες, δεν είναι μόνο τεχνολογικές οι καινοτομίες, αλλά και κοινωνικές. Ε, κάναμε και ε, θέματα καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας για τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, αλλά είναι και μεγάλος παράγοντας ε, ε, διαπολιτισμικού διαλόγου με τρίτες χώρες και θα θέλαμε αυτό το ευρωπαϊκό έτος να το προετοιμάσουμε ήδη από το 2017, να υπάρξουν κάποιες προκαταρκτικές και προπαρασκευαστικές διαδικασίες και συμμετοχή των κρατών μελών με μια λογική η οποία δεν θα είναι μόνο εθνική αλλά με προγράμματα και έργα τα οποία θα προωθήσουν την ευρωπαϊκή ε, διάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ε, και ε, της ηθαγένειας μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο συνάδελφος Διακόνου τώρα θα πάρει το λόγο, μετά θα σας πω λίγα πράγματα για το χρονοδιάγραμμα, το οποίο πρέπει να σεβαστούμε και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι επειδή όπως γνωρίζετε δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη και η Επιτροπή Προϋπολογισμών έδωσε συνέχεια στις τροπολογίες μας και τις έλαβε υπόψη, επομένως ε, η χρηματοδότηση για το ε, έτος πολιτιστικής κληρονομιάς ε, έχει ε, συμπεριληφθεί στον προπολογισμό εκτός ε, τη Δημιουργική Ευρώπη, που ήταν η αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εμεί θεωρούμε απαράδεκτη, διότι πάει να περικόψει ένα τομέα ο οποίο είναι ο τομέα που χρηματοδοτείται λιγότερο, ο του πολιτισμού. Να ευχαριστήσω λοιπόν και του συζητητέ και του κοιόδη συζητητέ τη Επιτροπή Πολιτισ... Ε, Προπολογισμών. Ο κύριος Δρογεύς και ο κύριος Μόργανο και άλλοι έδωσαν μάχη προκειμένου να καταφέρουν να δοθεί αυτό και να περάσει στου προπολογισμού και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή Προπολογισμών ε, αντιλαμβάνεται και την ανάγκη να υπάρχουν μεγαλύτερες δαπάνες για τον ε, πολιτισμό. Βέβαια, ελπίζουμε από εκεί και πέρα να τη τηρήσει και τη δέσμευση το Συμβούλιο, διότι πρέπει να υπάρχει προετοιμασία το 2017 και μετά έχουμε το Ευρωπαϊκό Έτος το 2018. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Διακόν για την παρουσίασή του. Ευχαριστώ. Ε, Uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ακολουθήσω τον ηρμό της σκέψης της Προέδρου, της κυρίας Κώστα, και να πω ότι πιστεύω ακραδάντως ότι αυτή η έκθεση είναι πραγματικά προϊόν συλλογικής εργασίας. Είναι μια έκθεση που ανήκει σε όλους μας. Εγώ βέβαια βάζω το όνομά μου από κάτω και υπογράφω, ωστόσο έχω συμπεριλάβει όλες τις ιδέες. Είναι ε, έκθεση της δικής μας Επιτροπής. Εάν λάβουμε υπόψη όλες τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα και διαβάσουμε την έκθεση, σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουμε. Είναι ένας φάκελος, μια υπόθεση που ακολουθεί την απλουστευμένη διαδικασία. Επομένως, οφείλουμε να σταθούμε σε πολύ συγκεκριμένες παρατηρήσεις και σχόλια και να κάνουμε το παν για να τα εφαρμόσουμε. Έχω κάποιες τροπολογίες να προτείνω, πολλά μπορεί να πει κανείς για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωστόσο θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρόλα αυτά γιατί ήταν πολύ πλήρης ο φάκελός της, πολύ πλήρες το κείμενο που παρουσίασε και δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιληφθεί ξεκάθαρα τον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως σας έλεγα όμως, η υπόθεση αυτή είναι πολύ περίπλοκη. Γνωρίζετε πολύ καλά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Γιούγκερ έχει ε, δώσει ένα τέλος στο προηγούμενο σύστημα των ευρωπαϊκών ετών κληρονομιάς. Και αυτή θα είναι η μόνη έκθεση που θα έχουμε κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας για το θέμα αυτό. Θα πρέπει ενδεχομένως να έχουμε στόχο να ε, αποκτήσουμε ένα συγκεκριμένο ρυθμό στη δράση μας. Δηλαδή, Μπορεί να καθυστερήσουμε, αλλά καλό είναι να μπει η έννοια της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ε, σε, σε, μια, σε ένα δρόμο και ελπίζω να μην είναι αυτό το τελευταίο έτος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Άλλωστε ελπίζω να είναι και το πιο ενδιαφέρον μέχρι σήμερα. Ε, είδα λίγο τι έχει γίνει τα προηγούμενα έτη, παρακολούθησα το πώς εξελίσσονται τα πράγματα και θεωρώ ότι δεν μπορούμε να υπερηφανευόμαστε για πολλές επιτυχίες. Δώσαμε έμφαση στην επικοινωνία, σε διασκέψεις, σε συνέδρια, σε τίποτα άλλο τελικά. Το βασικό θέμα είναι ο προϋπολογισμός το ποσό που μας προτείνουν είναι εξαιρετικά μικρό. Θα ζητήσουμε αύξηση του προϋπολογισμού και θα καθορίσουμε τα συγκεκριμένα ποσά που θα ζητήσουμε μαζί στην κοινή μας συζήτηση και θα βασιστούμε στους προϋπολογισμούς των παρελθόντων ετών. Ενδεχομένως να βγάλουμε το μεσοόρο των τελευταίων ετών και τελικά ίσως να καταλήξουμε στα 4 εκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση δεν συμφωνώ διό με το να δεν συμφωνώ με το ότι ο χρηματοδοτικός φάκελος για το 2018 έχει αφαιρεθεί από το πρόγραμμα ε, ε, Δημιουργική Ευρώπη. Εγώ, η κυρία Κώστα, ο κύριος Μαγκάνο έχουμε καταθέσει μια τροπολογία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά ενδεχομένως, και ζητούμε ε, ένα εκατομμύριο ευρώ περισσότερα για αυτή τη γραμμή του προπολογισμού και για προπαρασκευαστικές δράσεις. Άλλο σημαντικό θέμα είναι οι δραστηριότητε που προτείνονται για φέτος και θα ήθελα να έχουμε περισσότερες προτάσεις από εσάς και πιο γρήγορα κιόλα να υποβάλλετε προτάσεις. Το λέω γιατί πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι πρέπει να προχωρήσουμε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα θεωρώ ότι θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε περισσότερο τα κράτη-μέλη. Και αυτό προϋποθέτει πολλαπλασιασμό του προϋπολογισμού, γιατί κάθε χώρα μέλος έχει την υπερηφάνειά της και θα θέλει να ε, δώσει έμφαση και να προωθήσει τις δικές της αξίες τη δική της πολιτιστική κληρονομιά. Επομένως, χρειάζεται μεγαλύτερος προϋπολογισμός έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να δώσουν δείγματα της ε, κληρονομιάς τους, να δείξουν δηλαδή την κληρονομιά τους. Σας παρακαλώ λοιπόν, υποβάλλετε προτάσεις για δράσεις, για δραστηριότητα. Έχω πάρα πολλές ιδέες στο κεφάλι μου. Ε, βλέπω πάρα πολλές διεξόδους και ε, χρειάζομαι συνεργασία για να βρω λύση. Από εκεί και πέρα, ελπίζω να έχουμε τελικά και να μπορούμε να διανοηθούμε ευέλικτα σχήματα για τον προϋπολογισμό, να δημιουργήσουμε συνέργειες, να έχουμε συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, αλλά και συνέργειες με υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, να διασυνδέσουμε δηλαδή όλα αυτά και ίσως καταφέρουμε να αυξήσουμε το ε, τον προϋπολογισμό για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και μάλιστα κατά πολύ. Και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να εμπλέξουμε και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, τις αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Σε κάθε περίπτωση θέλω να συνεργαστώ με τη Γενική Διεύθυνση για την Επικοινωνία. Το έκανα αυτό Είδα τις δραστηριότητες των προηγουμένων ετών και είδα ότι πολύ μεγάλο μέρος των κονδυλίων κατευθύνεται στις δράσεις επικοινωνίας. Συμφωνώ, καλό πράγμα η επικοινωνία, να επικοινωνούμε τις δράσεις μας, αλλά δεν είναι αυτό ισορροπημένο. Υπερβολικά πολλά χρήματα παίρνει το σκέλος της επικοινωνίας. Θα πρέπει να μπορούν να καλυφθούν ορισμένα από τα ε, κόστη. Και έτσι θα μπορέσουμε εμείς να απελευθερωθούμε, να κάνουμε περισσότερα και να κινηθούμε καλύτερα φέτος. Πράγματι πρέπει να γίνουν εξοικονομήσεις, αλλά τουλάχιστον μια φορά στα πέντε χρόνια να έχουμε ένα έτος για την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό θέλουμε να, όταν μιλούμε για ρυθμό. Ε, δράσεων. Τουλάχιστον σε τακτά χρονικά διαστήματα να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Μία φορά στα πέντε χρόνια κοινοβουλευτική θητείας τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση ήθελα να πω και το εξή. Να προβλεφθούν κάποιες εκδηλώσεις σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης, σε ορισμένες περιοχές, εκθέσεις, ορισμένων συμβόλων εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε κράτους μέλους στον ίδιο χώρο, στην ίδια τοποθεσία. Έτσι θα αποκτήσει ορατότητα η ευρωπαϊκή διάσταση αυτού του εγχειρήματο. Αυτά λοιπόν, σας παρακαλώ να παρέμβετε, να επικοινωνήσετε μαζί μου, να διαβιβάσετε τις ιδέες σας, να συνεργαστούμε. Αύριο θα συναντηθώ με τους σκιώδεις εισηγητές, δεν ξέρω ακόμα τι ώρα. Και τέλος να πω ένα καλό νέο. που σχετίζεται με αυτά που είπα στην αρχή της παρέμβασής μου. Νομίζω ότι έχουμε κοινά στοιχεία όλες οι πολιτικές ομάδες, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Είναι κάτι που έχουμε από κοινού και μιλούμε για αύξηση του κατοφλίου των 5 εκατομμυρίων ευρώ για τα πολιτιστικά project, για τα πολιτιστικά προγράμματα και δράσεις και έργα χάρη στις κοινέ μας προσπάθειες ε, στο νέο δημοσιονομικό κανονισμό αυτό συμπεριλήφθη. Είναι ένα κείμενο το οποίο θα φτάσει σύντομα στην Ολομέλεια, θα φτάσει σύντομα στο Κοινοβούλιο. Μίλησα με τους αρμόδιους επιτρόπους πολιτισμού και ε, περιφερειακής ανάπτυξης και μου είπαν και οι δύο μου επιβεβαίωσαν ότι το ε, ανώτατο όρο των 5 εκατομμυρίων ευρώ δεν υπάρχει πια. Και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Για όλα τα υπόλοιπα αύριο θα έχουμε περισσότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και για το γεγονός ότι είστε διατεθειμένος να τίνετε δίκονους και να ε, συμμετέχει η Επιτροπή, ε, δεδομένου ότι υπάρχει και αυτή η ε, πιο ταχεία διαδικασία. Να πω επίσης ότι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ ενδιαφέρον και ε, με τη θεματολογία που θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι ε, πολύ συγκεκριμένα και υπάρχει αυτό που είπε και ο εισηγητής μας. Το 2017 ε, θα πρέπει να είναι μια χρονιά την οποία δεν θα πρέπει να χάσουμε. Θα πρέπει να είναι η χρονιά στην οποία θα καθορίσουμε την πορεία μας. Επομένως πρέπει να υπάρξουν προτάσεις ώστε ευθύ εξ αρχή να συμμετέχουν και τα κρατημέλη αλλά και ενδιαφερόμενοι για να δούμε τι δραστηριότητες θα χρειαστούμε εντό του 2017. Σας παρακαλώ να τηρήσετε τον χρόνο των τριών λεπτών, να δώσουμε το λόγο στους κοιόδης συγητές και μετά στους υπολείπους. Ο κύριος Δρογεύσκη. Mamy tu trzy zagadnienia i nie ich mieszać. Pierwsze zagadnienie to Πρόεδρε, Τρία θέματα έχουμε εδώ πέρα, τα οποία δεν θα πρέπει να συγχαίουμε μεταξύ μα. Ε, έχουμε ε, καταρχά ε, την έκθεση αυτή αυτή, τη οποία το κείμενο συζητάμε αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο είναι η χρηματοδότηση. Και το τρίτο είναι ο τρόπο ε, εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Έτου Πολιτιστική Κληρονομιά. Όσον αφορά το κείμενο, είναι αρκετά καλό ώστε να σας καλέσω να μην προτείνετε τροπολογίες. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Το κείμενο είναι καλό, δεν υπάρχουν επίμαχα σημεία, δεν έχουμε το χρόνο με το μέρος μας, πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Και θα ήθελα να ολοκληρώσουμε τις εργασίες εντός του χρόνου που έχουμε. Το δεύτερο θέμα είναι η χρηματοδότηση. όσο υψηλότερε είναι οι προσδοκίε μας, ε, τόσο καλύτερα θα πετύχουμε. Και είμαι πολύ ικανοποιημένο με το όσα έχει ήδη υιοθετήσει η Επιτροπή προπολογισμού. Προσπαθήσαμε να διασώσουμε τον προϋπολογισμό, αλλά από την άλλη αγωνιστήκαμε και για τα πιλωτικά μας προγράμματα και τα καταφέραμε. Από οικονομικής πλευράς λοιπόν είχαμε επιτυχία διότι το κατόφλι των 5 εκατομμυρίων ε, έγινε 10 εκατομμύρια, το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να συμπεριληφθούν και προγράμματα μεσαίου μεγέθους στις ε, πρωτοβουλίες ε, του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ανοιχτό προς παραμένει το τρίτο θέμα, το πώς θα τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Και πρέπει νομίζω να συζητήσουμε δύο συζητήσεις. Αυτό που ανέφερε η κυρία Τρούιπελ, ε, να εξετάσουμε τι θα γίνει με το 2019. Διότι θα πρέπει να συνοψίσουμε τις δράσεις και χρειαζόμαστε περισσότερα για το 2018. Και δεύτερη παρατήρηση, δεν επιτρέπεται να ξανασυμβεί αυτό που ήδη συνέβη, Το νέο πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Δημιουργικής Ευρώπης, ε, Creative Europe, το οποίο σημαίνει ότι παίρνουμε χρήματα από άλλα σημαντικά προγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή όλοι να έχουμε κατά νου ότι θα πρέπει να εγγυηθούμε την απαραίτητη χρηματοδότηση το 2018 και του χρόνου τον Ιούνιο. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην χάσουμε την ευκαιρία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις. Ο κύριος Μόργανο. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω. Ε, συμφωνώ με τα όσα ε, παρουσίασαν μέχρι τώρα οι συνάδελφοι. Σίγουρα πρέπει να ψηφίσουμε το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια την έκθεση αυτή. Ε, διότι αλλιώς θα χάσουμε χρόνο. Συγγνώμη, αλλά μικροφωνίζει ο ήχος. Ε, δεν θα προλάβουμε λοιπόν να τα καταφέρουμε γέρος. Ε, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να επαναλάβουμε κάποια πράγματα εδώ. Καταρχάν, το στόχο αυτού του ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να ε, αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, όσον αφορά την ιστορία, τις αξίες, την πολιτιστική κληρονομιά, να μάθουν για τον πλούτο της πολιτιστικής ποικιλομορφία ως ένα εργαλείο για να μπορέσουν να αυξήσουν την αίσθηση της ηθαγένειας, του ανήκειν. Ε, επίσης, πρέπει να υπάρχει και μια προοπτική για το μέλλον, ε, την οποία θα πρέπει να προωθήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα πάντα ε, δεν θα πρέπει ε, να είναι μια αυτό εκτίμηση για τα ε, επιτεύγματά μας. Όπως είπε και ο πρόεδρος και η πρόεδρος και ο εισηγητής υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες τις οποίες βεβαίως πρέπει να εμπαθύνουμε. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα σήμερα το πρωί αλλά πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε συνέχεια σε αυτές τις πρωτοβουλίες στη διάρκεια του έτους. Δηλαδή για να σηματοδοτήσουμε καταλήλως τα πράγματα αυτά πρέπει να υπάρχει ένα λογότυπο, ε, ε, ένα, μια ονομασία η οποία θα ε, δίδει αξία σε αυτό τον εορτασμό. Ε, δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα μόνο σε επίπεδο ένωση. Πρέπει να υπάρχει πραγματική συνεργασία και από πλευρά κρατών μελών και θα πρέπει λοιπόν εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προτρέψουμε τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίω από την πλευρά τη ε, να ε, συμμετέχουν ουσιαστικά, να συμμετέχουν τα διάφορα επίπεδα αν θέλουμε πραγματικά να φτάσουμε και στο υψηλότερο επίπεδο, πρέπει να υπάρχει συμμετοχή και σε εθνικό και σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, διότι αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να φτάσουν πραγματικά στους ανθρώπους που είναι τελικά ο στόχος αυτής της δράσης. Εδώ Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και ε, σωστή σχέση δημοσίου ιδιωτικού τομέα, δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα επιλύσουμε. Εμείς υποστηρίζουμε μια νέα γραμμή προϋπολογισμού σαφέστατα στο θέμα αυτό. Να μην ενταχθεί ε, το ζήτημα στην ε, χρηματοδότηση της Δημιουργικής Ευρώπης. Βεβαίως θα πρέπει να προσθέσω ότι κατά την άποψή μου θα μπορούσαμε να υποφεληθούμε και από κάποιες ε, χρηματοδοτήσεις ε, που προκύπτουν από την εγκάρσια προσέγγιση μεταξύ των γενικών διευθύνσεων που θα είναι αρμόδιες για το ευρωπαϊκό έτος. Δεν είναι μία η γενική διεύθυνση και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι και σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να ε, έχουμε κάποια πρόσθετα στοιχεία. Θα ήθελα να προσθέσω και μία πτυχή την οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, να ενισχύσουμε και την διοργανική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παραδείγματος χάρη, ε, δεν υπάρχει συγκεκριμένη συγκεκριμένη παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στο έγγραφο υπάρχει μια συγκεκριμένη αναφορά στο άρθρο 5 του σχεδίου απόφασης, το οποίο είναι ακόμα προς συζήτηση, και προβλέπεται να υπάρχουν εθνικοί συντονιστές ε, και ε, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να υπάρχει και παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να δώσουμε και μία κατεύθυνση, γιατί εμείς επιμένουμε στο έτος αυτό και βεβαίως ε, δεν ε, ε, είναι δυνατόν να επιληθούν τα πάντα το 2018. Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις προτάσεις. Ο κύριος Λιουερ δεν εδώ. Ο κύριος Μαλτέζη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι ιδέες και προτάσεις εξαρτώνται και από τη χρηματοδότηση και η χρηματοδότηση είναι πενιχρή. Επειδή βεβαίως Πάντα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εγώ θα ήθελα να βρούμε έναν τρόπο για να απαντήσουμε λίγο πιο ε, ριζοσπαστικά στο γεγονός ότι δεν επενδύουμε στον πολιτισμό. Διότι αναφερόμαστε στο έτος πολιτιστικής κληρονομιάς, ε, ένα από τα πιο σημαντικά ε, στοιχεία, πηγή πλούτου. Αν συζητούσαμε για τη χρονιά του Μερλούκιου θα παίρναμε πολύ περισσότερα χρήματα. Όσο και αν μ' αρέσει ο Μερλούκιος ως ψάρι νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να επενδύουμε μόνο σε αυτό. Μεταξύ των προτάσεων υπάρχουν κάποιες πάρα πολύ χρήσιμες. Ε, μία από αυτές ε, τι παρουσίασε ο εισηγητής ε, αυτή την ενιαία θηρίδα, αυτό το, τη διαδικτυακή πύλη. θεωρώ ότι είναι μία πολύ καλή πρόταση και κυρίως πολύ χρήσιμη. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξεκινήσει και μπορεί να έχει πολύ καλή σύνδεση. Τώρα, επειδή ακριβώς δεν είναι πολλά τα κονδύλια, θα πρέπει να ε, επικεντρωθούμε, να έχουμε ένα λογότυπο, αλλά και ένα στόχο. Παραδείγματος χάρη, η πρόταση να απευθυνθούμε στους νέους. Εγώ θα ήθελα να προτείνω και ε, ε, να ε, τονίσουμε και πόσο ευάλωτη είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά και πόσο γίνεται όλο ένα και πιο ευάλωτη. Διότι ε, κάποιες από τις χώρες μας, για παράδειγμα, λόγω περικοπών των δημοσίων προγραμμάτων ή λόγω κλιματικών αλλαγών ή λόγω φυσικών καταστροφών, η πολιτιστική κληρονομιά σε όλη την Ευρώπη, δυστυχώς και κυρίως στις πιο φτωχές χώρες, ε, είναι όλο και πιο ευάλωτοι. Και αυτό είναι ένα ακόμα από τα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τρούπελ. Yes, thank you, Ευχαριστώ, Σίλβια. Εγώ νομίζω ότι τώρα όταν συζητάμε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και γενικότερα την έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό να καταστήσουμε σαφές ε, ποια κατανόηση του πολιτισμού επιδιώκουμε και νομίζω ότι θέλουμε περισσότερο δημοκρατική δημοκρατικό πολιτισμό και να μην θεωρούμε ότι ένας πολιτισμός είναι ανώτερος από κάποιον άλλον, διότι έχουμε πολύ πικρές εμπειρίες ε, στην Ευρώπη ε, σχετικά με ε, την έννοια του πολιτισμού, όπου ένας πολιτισμός θεωρείται ανώτερος από κάποιον άλλον. Εάν τονίσουμε λοιπόν τον εθνικό πολιτισμό, αυτό μάλλον διαιρεί τον κόσμο. Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι θα ξεκινήσουμε με βάση τον δημοκρατικό πολιτισμό και την ε, ένταξη της συμμετοχικότητα. Και αν υπάρχουν ε, μειονότητες να είναι ανοιχτές ε, και να υπάρχει πολιτικό σκηνικό για την πολυμορφία. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την κατανόηση του δημοκρατικού πολιτισμού και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι η έννοια που θα μας καθοδηγεί κατά τον εορτασμό της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτήν την ε, τεράστια πολιτική συζήτηση σχετικά με το αν μπορούμε να συνεπάρξουμε με διάφορες μειονότητες ε, και θρησκείες. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δείξουμε ότι δεν έχουμε σχέση με τρομοκράτες και εχθρικές δραστηριότητες, αλλά ότι πρέπει να υπερασπιστούμε αυτήν την ανοιχτή κοινωνία. Γι' αυτό είναι σημαντικό στην έκθεση αυτή να συνεργαστούμε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να συμμετάσχουν πολλοί και να μην περιοριστούμε μόνο σε κάποιους φορείς. Αλλά να είναι μια ανοιχτή εκδήλωση για το σύνολο της κοινωνίας. Και τελευταία μου παρατήρηση, θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο συνάδελφος. Χρειαζόμαστε νέα γραμμή του προπολογισμού. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στο πλαίσιο ε, του προγράμματο Δημιουργική Ευρώπη, διότι είναι υπερβολικά περιορισμένο το πρόγραμμα αυτό για τη συγκεκριμένη χρήση. Και θα πρέπει να βρούμε συμμάχους ε, στο Κοινοβούλιο και να καταστήσουμε σαφές ότι το θέμα δεν είναι αυτό το περιορισμένο πρόγραμμα της ε, δημιουργικής του δημιουργικού πολιτισμού είναι ένα θέμα που ε, αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε επιπλέον πόρους και να δημιουργήσουμε νέα γραμμή του προϋπολογισμού. Σύμφωνα απολύτως, η κυρία Αντινόλφη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ στα δελτία τύπου διαβάζω εξαιρετικά πράγματα για αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ε, πριν ε, διάβαζα να προωθήσουμε τη συνειδητοποίηση ε, μιας ιστορίας και μιας κοινή ταυτότητας, βοηθά τη συνοχή, την κοινωνική ένταξη μέσω αναβάθμισης και υποβαθμισμένων περιοχών. Πολύ ωραία πράγματα όλα αυτά. Εμείς μπορεί να μιλάμε βέβαια για πολιτιστική κληρονομιά, άειλη, όπως έλεγε ο Κούρτσιο Μαλτένριζε, αλλά και για ε, ηλική ε, πολιτιστική κληρονομιά. Αλλά το πρόβλημα είναι κοινό. Εάν δεν υπάρχει ένας ελάχιστος ε, προϋπολογισμός, ε, θα είναι πολύ αδύναμη αυτή η εικόνα που θα παρουσιάσουμε και ελοχεύει και ο κίνδυνος να μην ενταληφθούν καν οι πολίτες ότι υπάρχει Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής κληρονομιά. Είναι λοιπόν σαφές ότι εάν δεν υπάρχει κατάλληλη γραμμή προϋπολογισμού, αξιοπρεπής και εμείς από πλευράς μας βεβαίως θα δεσμευθούμε ώστε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις ε, για να μπορέσουμε να έχουμε ε, και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος εντό εισαγωγικών ε, να ε, σταθούμε λοιπόν σε δράσεις ε, συγκεκριμένες ε, και σε πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να έχουν συγκεκριμένη προβολή ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε μια πολύ άσχημη εικόνα και τελικά να μην μπούμε στους πολίτες αυτό που προσπαθούμε να πούμε. Δηλαδή αντί να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά τους λέμε να, ορίστε, βγάζουμε μια ωραία εικόνα και λέμε ότι αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής και στην πραγματικότητα δεν επενδύουμε σε τίποτα γιατί δεν το πιστεύουμε. Ε, δεν πρέπει λοιπόν να πέσουμε σε αυτή την παγίδα και πέραν τη ε, ε, ε, άποψης που έχει κάθε πολιτική ομάδα, θα πρέπει όλοι από κοινού να προσπαθήσουμε να πετύχουμε έναν αξιοπρεπή προπολογισμό. Ευχαριστώ. Έγινε η προσπάθεια στην Επιτροπή Προπολογισμών βεβαίω, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε για να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση και του Συμβουλίου. Η κυρία Μπίλντε δεν θέλει το λόγο. Α, είστε σκιώδη συγγήτρια και νόμιζα ότι θα θέλετε το λόγο. Όχι. Η κυρία Πόξερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ε, βρίσκω πολύ καλή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν πάνω στο θέμα αυτό, ότι είναι σημαντικό θέμα δηλαδή το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και νομίζω ότι υπάρχει συνένεση όχι μόνο μεταξύ των πολιτικών ομάδων, αλλά και μεταξύ των κρατών μελών, διότι είναι θέμα σημαντικό για όλους μας. Κάθε κράτος μέλος έχει πολιτιστική κληρονομιά που θέλει να δείξει και να διατηρήσει. και που θέλει να αναδείξει και εντός ε, της χώρας ε, και ε, στις γειτονικές χώρες. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι σημαντικό, διότι έτσι μπορούμε να επιστρέψουμε στις ρίζες της Ευρώπης. Εάν σκεφτούμε όμως το θέμα της νεολαίας, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι στον τομέα της πολιτικής κληρονομίας απασχολούνται πάνω από 300.000 ε, άτομα. Ε, αν ε, λοιπόν επιτύχει το εγχείρημα αυτό και πραγματοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης στον τουρισμό, σε υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνίες και σε πολλούς άλλους τομείς. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε σίγουρα αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Äh, Ο κύριος Κόσνερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω λίγα λόγια σχετικά με την πραγματοποίηση αυτής της ιδέας. Η Ευρώπη ως πολιτιστικός χώρος ε, σίγουρα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά ώστε οι πολίτες ε, να αποκτήσουν κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση. Και γι' αυτό χαίρομαι με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το Ευρωπαϊκό Έτος πολιτιστική Κληρονομιάς. Η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει κοινή πηγή πολυμορφίας και δημιουργικότητας ε, και να ε, δείξουμε και πόσο σημαντικά είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό θέλω να συμφωνήσω με τη συνάδελφο την Χέλγα Τρίπελ. Πιστεύω λοιπόν ότι ένα τέτοιο ευρωπαϊκό έτος μπορεί να συμβάλλει στην ε, ε, αντιμετώπιση του αναδυόμενου εθνικισμού στα κράτη-μέλη. Σημαντικό επίσης είναι να έχουμε κατά νου την προώθηση της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Εγώ προέρχομαι από την περιοχή Ρουρ και έχει πολύ σημαντική... έχει πολύ μεγάλη σημασία η βιομηχανία στον τομέα αυτών για τη ζωή των πολιτών. Και σε άλλα μέρη της Ευρώπης ε, βλέπουμε αναβίωση παλαιών βιομηχανικών χώρων. που συμβάλλουν σημαντικά και για τη μεταρρύθμιση στην Ευρώπη. Οι πολίτες στην Πολωνία, την Ουγγαρία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε άλλες περιφέρειες, βλέπουν πώς ε, με την ε, ιδιοποίηση ε, βιομηχανιών που είχαν παροπλιστεί δημιουργείται κέρδος για τις περιοχές αυτές. Και οι άνθρωποι που έχουν ζήσει εκεί και που έχουν αγωνιστεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να τους ε, θυμόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ε, κοινωνικά προγράμματα και γι' αυτό θεωρώ σημαντικό στο έτος αυτό να αποτελέσει μέρος ε, του έτους αυτού η ο αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις περιοχές αυτές, διότι ε, σε πολλά μέρη της Ευρώπης ε, έχουν αγωνιστεί οι άνθρωποι για τα εργατικά δικαιώματα από τα οποία υποφελούμαστε όλους. Μπορούμε λοιπόν όλοι να μάθουμε από τη διαδικασία αυτή. Μπορούμε να μάθουμε ότι η κοινωνική πρόοδος δεν έρχεται από μόνη της, πρέπει να αγωνιστεί κανείς για αυτήν και κάθε πτυχή αυτού του θέματος ε, θα πρέπει να βρίσκεται στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού έτους. Η ανάπτυξη λοιπόν ε, ε, της βιομηχανίας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της πολιτιστικής κοινωνίας της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Μου άρεσε η ιδέα του κυρίου Διακόνο να συμπεριληφθούν δηλαδή όλα τα κράτη-μέλη στο ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς. Όμως ο κύριος Μοργάνο πήγε πέρα και λέει να συμπεριλάβουμε και τοπικές και περιφερειακές αρχές. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους νέους. Να ξεκινήσουμε ένα διαγωνισμό για τους νέους, για το ποιο θα είναι το κόνσεπτ για την κήρυξη του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Για το Ευρωπαϊκό Έτος Αθλημάτων το σλόγγαν το σκέφτηκε ένα 12χρονο παιδί. Απευθύνω λοιπόν κάλεσμα να ακούσουμε περισσότερο τους νέους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φερχάιγεν. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε πολύ καλέ ιδέε σχετικά με το πώ μπορούμε να διαμορφώσουμε το ευρωπαϊκό έτο πολιτιστική κληρονομιά. Ένα όμω θα πρέπει να είναι σαφέ. Επιτυχία θα αποτελέσει μόνο εάν τα κράτη-μέλη, οι περιφέρειε, οι δήμοι, ε, οι πολιτιστικέ ε, πόλει ε, συνεργαστούν και στην διοργάνωση. Εάν εμείς από πάνω ως Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλουμε κάτι, τότε το αποτέλεσμα μετά από ένα χρόνο θα ξεχαστεί. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν όλοι και να δημιουργήσουμε δίκτυα. Διότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέλουμε να καταπολεμήσουμε ε, τα εθνικιστικά κινήματα και ακριβώς ε, στον αγώνα αυτών μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο ε, οι εκδηλώσεις για την πολιτιστική κληρονομιά. Θα πρέπει να δούμε τι κοινό έχουμε, πού υπάρχουν παράλληλες εξελίξεις, ποια είναι η κοινή μας πορεία και ποιε είναι οι υποχρεώσεις μας για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτή είναι η προστιθέμενη αξία που μπορούμε ε, να αποκομίσουμε από το έτο αυτό όσον αφορά τον προϋπολογισμό που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, οι προσδοκίες ε, είναι υψηλές. Δεν θα μπορέσουμε να ανακαινήσουμε όλους τους ε, πολιτιστικούς ε, χώρους. Ε, νομίζω ότι πολλοί κόσμος δεν έχει καταλάβει ποιος είναι ο στόχος ενός τέτοιου έτους. Στόχος του έτους αυτού είναι να ξεκινήσουν συνεργασίες, να ξεκινήσουν πρωτοβουλίες. Θα πρέπει λοιπόν με λογικό και φρόνιμο τρόπο να φροντίσουμε να συμμετάσχουν όλα τα κράτη-μέλη ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα βιώσιμο. Ευχαριστώ. Κυρία Καμερέβερτη, είναι πολύ ε, σημαντικό αυτό το θέμα της βιωσιμότητας που μόλις ε, αναφέρθηκε. Όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες ε, και τον ρόλο τους, έχουμε τονίσει ότι θα πρέπει να είναι βιώσιμες οι προτάσεις και όχι απλά να προωθήσουμε μία ελίτ του πολιτισμού, αλλά με τον θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσες, αλλά και με ένα τέτοιο ευρωπαϊκό έτος της πολιτιστικής κληρονομιάς, να συμμετάσχουν οι πολίτες. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν ε, τοπικές και περιφερειακές επαφές. Ε, η κυρία Κώστερ είπε ότι δεν μιλάμε εδώ για ε, πολιτιστική ελίτ, ε, συναυλίες, ε, θεατρικές παραστάσεις, και κλασικά μνημεία. Δεν είναι ακριβώς ε, αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως ε, ο μη υλικός ε, πολιτισμός, οι παραδόσεις που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Και να γίνουν κατανοητέ αυτέ οι παραδοσει ε, όχι ως διάκριση από άλλους, ε, κάτι διαχωριστικό από άλλους, ε, αλλά κάτι που μας ενώνει. Να μην λέμε δηλαδή ότι η δική μου παράδοση είναι καλύτερη από τη δική σου, αλλά να προσπαθήσουμε να υπάρξει και πολιτιστική κατανόηση και συνεννόηση και στον άειλο πολιτισμό. Τα μη υλικά πολιτιστικά αγαθά μπορούμε να τα επιβάλλουμε αυτά από πάνω, μπορούμε να προτείνουμε κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ε, τα κράτη-μέλη, αλλά τα κράτη-μέλη, και εδώ έχουμε όλοι να παίξουμε ένα ρόλο, να φροντίσουμε να εφαρμοστεί η ιδέα αυτή. Ότι δεν θέλουμε απλά ελιτιστικό πολιτισμό, Θέλουμε ένα έτος όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες να σκεφτούν την ιστορία τους και να σκεφτούν και το μέλλον τους ε, με ε, ανταλλαγές ε, απόψεων και ιδεών. Ευχαριστώ. Η Julie Ward. Ευχαριστώ πολύ συναρπαστική συζήτηση και συμφωνώ με πολλούς από τους προλαλήσαντες, ειδικά στο να εμπλέξουμε τους νέους. Πράγματι, οι νέοι θα διαμορφώσουν το μέλλον όλων μας και είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα σε όλα τα επίπεδα. Είναι εξαιρετικά, ε, εξαιρετική ευκαιρία να δείξουμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι κάτι το άκαμπτο και ότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι ένα πλούσιο μείγμα διαφορετικών εθνοτήτων, γλώσσεων, θρησκευτικών ε, δογμάτων, κυμάτων μετανάστευσης και προσφύγων, αλλαγών μετακινήσεων. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ευρώπη είναι κάτι που συνέβαινε πάντοτε ε, εδώ και αιώνες. Έχουμε πρόσφυγες ουγενότους που ήταν στις απαρχές της δικής μου πολιτιστικής κληρονομιάς. Ε, ήρθαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και έφεραν το εμπόριο ε, των υφασμάτων, της δαντέλας. Και η πόλη που γεννήθηκε ο πατέρας μου πλούτησε χάρη στην τεχνογνωσία ε, της δαντέλας που έφεραν οι ουγενότοι πρόσφυγες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι καινούριο αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα με τους πρόσφυγες στην Ευρώπη και είναι κάτι που πρέπει να είναι εξαιρετική ευκαιρία να γιορτάσουμε τη διαφορετικότητα, την πολυμορφία και να γιορτάσουμε την μετανάστευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ, Έχουμε τον ε, κύριο Τζαμπιέρη, τμήματάρχη του ε, τμήματος ε, για τον πολιτισμό και την κυρία Τσακιτάνο που είναι μαζί του, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Ε, μετά θα σας πω το χρονοδιάγραμμά μας ε, στο τέλος. Αλλά τρεις ε, παρατηρήσεις. Να πω ότι συμφωνώ απολύτως ότι το έτος αυτό πρέπει να αποδείξει ότι είναι το ευρωπαϊκό έτος ε, πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και της ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Να έχει δηλαδή μια ισχυρή διεθνή διάσταση ε, και, για να λάβουμε υπόψη καταρχάς το θέμα της ταυτότητας και ε, επίσης και τις πρωτοβουλίες και τα δίκτυα τα οποία υπάρχουν ήδη. Υπάρχουν πολύ σημαντικά δίκτυα. Η, πολιτιστικές πρωτεύουσες για παράδειγμα, ε, τα πολιτιστικά δίκτυα τα οποία ήδη ε, ε, υπάρχουν και επίσης μία σχέση με αυτό που είπαμε, δηλαδή οπτικοακουστικά θέματα, άειλα και υλικά πολιτιστικά αγαθά. Επίσης, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, κάποιος το είπε και θα ήθελα να ακούσω και κάποια απάντηση, τουλάχιστον για το κατά πόσο είναι διατεθειμένη να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα λογότυπο, ε, ε, ένα όνομα, μία μάρκα και μία δικτυακή πύλη. Έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα ε, μήνυμα ότι υπάρχει ένα κατάλληλο πλαίσιο, να συμμετέχει τρίτον και η περιφερειακή και η τοπική κοινωνία στις δραστηριότητες αυτό ε, είπε ο κύριος Διακόνου και οι συνάδελφοι ότι η διακυβέρνηση όπως προβλέπεται πρέπει να προβλέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι σημαντικό, νομίζω ότι γίνεται γενικότερα στο Ευρωπαϊκό έτος. Κάθε χώρα έχει και συγκεκριμένη ε, διακυβέρνηση και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να συμμετέχουν και οι νέοι και με κάποιες... Ε, δραστηριότητες υπέρ της δράσης και για τι ε, γνώσεις, αλλά στην Ιταλία υπάρχει και για παράδειγμα ένα ε, παράδειγμα που λέγεται «Υιοθέτησε ένα μνημείο». Ε, είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και δείχνει και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να προωθήσουμε και τον πολυπολιτισμικό διάλογο, να γνωρίζουμε και τις διάφορες πολιτιστικές πραγματικότητες και κάτι ακόμα. Για το 2017 δικαίως ε, βλέπω ότι θέλουμε να δώσουμε περιθώριο πέραν στο θέματα του προπολογισμού και στην ε, προετοιμασία και την ενεργή συμμετοχή των κρατών μελών, των ενδιαφερομένων ε, για να υπάρχει επικοινωνία και να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε. Ίσως, και επιτρέψτε μου να κάνω εδώ μια μικρή πρόταση που προέκυψε και από την ομάδα σκέψης που δημιούργησαν για την πολιτιστική πληρονομιά αρκετά κρατημέλη και με την οποία είχαμε επαφές, γιατί να μην έχουμε το 2017 και κάποιες θεματικές εκδηλώσεις για το ε, έτος πολιτιστικής κληρονομιάς που θα γίνουν σε ε, εμβληματικά μνημεία ε, να προετοιμάσουμε δηλαδή ε, λίγο το θεματολόγιο και να ε, τονίσουμε τους στόχους μέσω κάποιων εκδηλώσεων, οι οποίες σαφέστατα πρέπει να συγχρηματοδοτηθούν και από τα κράτη-μέλη και με, από ιδιωτικούς εταίρους ίσως, αλλά να είναι μια μορφή παρουσίασης και ε, έγκαιρης ε, συμμετοχή συμμετοχής, αυτό το έτος που θέλουμε να έχει μεγάλη συμμετοχή. Ε, συγγνώμη, ήθελα να κάνω κι εγώ κάποιες παρατηρήσεις για να βοηθήσω ίσως και εγώ τις εργασίες του συναδέλφου Διακόνου. Να δώσω αμέσως τώρα το λόγο στον κύριο Τζαμπιέρη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μια πολύ σημαντική πρόταση για εμάς, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ευχαριστώ ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την δική σας Επιτροπή γιατί δούλεψα, δουλέψατε πάρα πολύ σκληρά να μπορέσει να υπάρξει και να προωθηθεί η πρόταση αυτή. Και η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, ομολογώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω εν συντομία το δικό μας κόνσεπτ, η δική μας αντίληψη, γιατί το προτείναμε το έργο αυτό με τον τρόπο που το προτείναμε. Θέλαμε η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά να ενταχθεί σε μια ευρύτερη διαδρομή και γι' αυτό το συνδέσαμε με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον πολιτισμό και υπενθυμίσαμε όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, γιατί θεωρούμε ότι αυτός ο, ο χρόνος είναι ένα έτος ε, που είναι ευκαιρία για την παγίωση των κεκτημένων και για την επιτάχυνση του ρυθμού των δράσεών μας. Και γι' αυτό η διάσταση mainstreaming είναι απαραίτητη, είναι ουσιαστική. Τότε δηλαδή πολλά τμήματα και διαφορετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκής Επιτροπής ασχολούνται με αυτό το θέμα. Το mainstream είναι απαραίτητο γιατί ε, υπάρχουν κονδύλια για την πολιτιστική ε, κληρονομιά τα οποία διαχειρίζονται και διοχετεύουν άλλα τμήματα και άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, π.χ. τα διαρθρωτικά ταμεία μεταξύ άλλων που 6 δις ευρώ διαχειρίζονται από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές με αντικείμενο την πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχουν λοιπόν κονδύλια και πολύ σημαντικά. Και το mainstreaming επίσης είναι σημαντικό για την ε, κληρονομιά που θα αφήσουμε πίσω, πίσω μας. Δεν είναι μια και έξω. Είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη των, ε, των πολιτικών μας και έρχεται την κατάλληλη στιγμή όπου θα ζητούμε τη μελλοντική γενιά προγραμμάτων και γι' αυτό είναι σημαντικό να το κάνουμε σωστά. Συμφωνούμε με όλα όσα υπόθηκαν για την κοινωνική διάσταση και κυρίως την ευρωπαϊκή διάσταση. Σήμερα έχουμε σημαντικά κονδυλία και είναι διαθέσιμα σε ε, κρατικό επίπεδο. Επομένως, το ευρωπαϊκό έτος έχει σαν στόχο να φωτίσει την ευρωπαϊκή διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μία κληρονομιά που διαμορφώθηκε σε βάθος χρόνου, αλλά και από το ένα σύνορο στο άλλο, ε, ανεξαρτήτως σύνορων. Και αυτό είναι μια κληρονομιά κοινή που έχουμε και σχετίζεται και με το ψήφισμα που παρουσιάστηκε και είναι απολύτως απαραίτητο αυτό το κριτήριο και αυτός θα πρέπει να είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έννοια της δημοκρατικής ε, κουλτούρας και της ανοιχτής κοινωνίας είναι απολύτως απαραίτητη. Ε, αυτή τη δουλειά κάνουμε με τα κράτη-μέλη, την συμμετοχική διακυβέρνηση για να δούμε πώς διαχειριζόμαστε τις κληρονομιά, ε, την κληρονομιά μας. Δεν θέλουμε απλά προθήκες και βιτρίνες, θέλουμε να αφήσουμε κληρονομιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε όλα τα τμήματα, σε όλες τις υπηρεσίες, να υπάρχει συμματοχική διακυβέρνηση, ε, ε, να υπάρχει αυτή η διάσταση για τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και είναι και ευκαιρία να φωτίσουμε και το ρόλο της εκπαίδευσης για την πολιτιστική κληρονομιά. Σαφέστατα, ε, βασικοί συνομιλητές μας είναι οι νέοι και θα κινητοποιήσουμε και όλα τα άλλα εργαλεία. Η κυρία Κώστα άλλωστε σας υπενθυμίσε ότι έχουμε δίκτυα, υπάρχει δουλειά που έχει γίνει. Έχουμε τα βραβεία, έχουμε τα ευρωπαϊκέ ημέρε πολιτιστική κληρονομιά που διαχειριζόμαστε από κοινού με το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Όλα αυτά είναι εξαιρετικέ ευκαιρίε. Μπορούμε να κινητοποιήσουμε όλα αυτά που έχουμε στη διάθεσή μα. Και βεβαίω δεν έχουμε αντίρρηση για υψηλότερο προπολογισμό. Αυτό είναι αυτονόητο. Σε va sans λένε οι Άγγλοι. Οι Γάλλοι, με συγχωρείτε. Και λέει ο μιλητής, και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε μια αξιοπρεπή δουλειά. Ε, να υπενθυμίσουμε ότι Το Creating Europe, η δημιουργία της Ευρώπης, είναι σημαντικό για εμάς για δύο λόγους. Πρώτον, διότι προωθεί την ευρωπαϊκή διάσταση και δεύτερον, συνδέεται με, ε, με τη βιομηχανία του πολιτισμού και του τουρισμού. Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, έστω και ανεξάρτητα, και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τέλος, Ως προς την ε, συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην συμμετοχική διακυβέρνηση δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Το λόγο, το, ε, η ονομασία, η διαδικτυακή πύλη, όλα αυτά τα δουλεύουμε τώρα, είναι σημαντικά είναι σημαντικά γιατί ποτέ δεν θα έχουμε αρκετά χρήματα να γίνουν πρωτοβουλίες σε όλα τα κράτη-μέλη που να απευθύνονται σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Βεβαίως χρειαζόμαστε τη βοήθεια των κρατών μελών και θα μπορέσουμε να κατονομάσουμε ε, πρωτοβουλίες ε, για να έχουν μεγαλύτερο βελινεκές και να τις διαδώσουμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ όμως για το όραμά σας, το οποίο συμμερίζεται πλήρως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις και για το γεγονός ότι είστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε. Να πω το εξής, εγώ δεν πιστεύω ότι η δημιουργική Ευρώπη ε, θα πρέπει να συνδυαστεί ε, με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ε, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι οι πόροι. Πρέπει να υπάρξει μια καλή συμμαχία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Ο εισηγητής τώρα, παρακαλώ. Ε, ε, προκειμένου να υπάρχει επιτυχία σε αυτά τα προγράμματα, ε, πρέπει αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς να είναι διαφορετικό από όλα τα διάφορα ευρωπαϊκά έτη για οτιδήποτε. Διότι αλλιώς ε, θα είναι μονότονα τα πράγματα και απλώς θα κάνουμε τα ίδια με κάθε χρονιά από την ε, σημερινή συζήτηση διαπιστώσαμε ότι τα θέματα αυτά πρέπει να είναι απόλυτα σαφή. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της κληρονομιάς. Επιμένω ως προς τον όρο χαρακτήρας και πρέπει να αντιληφθούμε γιατί ο πολιτισμός ε, μας αφορά όλους. Χρειαζόμαστε λοιπόν να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή εθνικισμού η οποία μας οδηγεί σε πράγματα τα οποία δεν επιθυμούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και πρέπει να σας πω ότι με πόνεσε το χέρι μου από όλες τις σημειώσεις που κράτησα για να σημειώσω όλα αυτά τα οποία είπατε διότι τα πάντα έπρεπε να ε, καταγραφούν και θα τα πούμε στη συνέχεια. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές προτάσεις ζήτησες από τους συναδέλφους ε, να σου κάνουν προτάσεις και όλοι έκαναν προτάσεις. Θα ήθελα απλώ να υπενθυμίσω ότι μετά από αυτή την ανταλλαγή απόψεων το τελικό σχέδιο του ε, του κειμένου με τι τροπολογίε που θα συζητηθούν μεταξύ των εισηγητή, του εισηγητή και των σχεδόν εισηγητών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τι 14 Οκτωβρίου και θα δοθεί ε, από την υποφαινόμενη στα μέλη τη επιτροπή Πολιτισμού. Μετά από εκεί και πέρα έχουν 21 μέρε τα μέλη για να πούν αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Εάν πάνω από το 10% δηλαδή εάν πάνω από 4 μέλη τη Επιτροπή διαφωνούν τότε θα πρέπει να περάσουμε σε ψηφοφορία. Η ψηφοφορία σε περίπτωση που πρέπει να γίνει θα γίνει στι 8 Νοεμβρίου Νοεμβρίου ή στις 28 Νοεμβρίου. Αλλά όχι για να κατατεθούν νέε τροπολογίε, αλλά μόνο για να ψηφίσουμε αυτές οι οποίες ε, πρότεινε ο εισηγητής. Αυτή είναι η απλουστευμένη διαδικασία. Εάν όμως δεν υπάρχουν ενστάσεις, η έκθεση θεωρείται ότι εγκρίνεται και θα πάει απευθεία στην Ολομέλεια. Ε, όπου και θα ψηφιστεί το Δεκέμβριο του 2016. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να ε, ψηφίσουμε και το Νοέμβριο, θα προσπαθήσουμε βεβαίως, αλλά πρέπει να ψηφιστεί μέχρι το Δεκέμβριο. Αυτά λοιπόν, ε, να ευχηθώ καλή δουλειά στον εισηγητή και στους κοιόδης εισηγητές. Είμαι βέβαιος ότι, βέβαιη συγγνώμη, ότι θα υπάρξει μια πολύ καλή παρουσίαση και ε, όλοι οι συνάδελφοι που θέλουν να συνεργαστούν, καλό είναι να έρθουν σε επαφή με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητής μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να περάσω σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την Επιτροπή μας, την παρουσίαση των νικητών του ε, βραβείου νέων Καρλομάγνος. Είναι ήδη εδώ άλλωστε οι νικητές. Πρόκειται για μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, τη γνωρίζετε. Το βραβείο Καρλομάγνου θεσπίστηκε το 2008 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το Διεθνές Ίδρυμα για το βραβείο Καρλομάγνου του Ακουής και βραβεύει ε, νέους, όπως σας είπα, θα ακούσουμε και την άποψή τους βεβαίως γι' αυτό. Βραβεύει λοιπόν νέους που ε, υπέβαλαν ε, προγράμματα. Παρακαλώ, καλώς ορίσατε, καθίστε. νέους που ε, προώθησαν προγράμματα τα οποία προωθούν ε, την ανάπτυξη μιας κοινή αίσθηση ταυτότητας και ευρωπαϊκής συνειδητοποίησης μεταξύ των νέων και προτείνουν συγκεκριμένα παραδείγματα Ευρωπαίων πολιτών που συμβιώνουν σε μια κοινότητα. Οι νέοι που έχουμε εδώ και σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλωσορίσατε λοιπόν. και εκ μέρους των ε, μελών της Επιτροπής και χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Ε, συγχαρητήρια και για τις ε, ε, νίκες σας και έρχομαι εδώ λοιπόν στα αριστερά μου. Το νικητή του πρώτου βραβείου είναι το Integrate από την Ιταλία. Εχθές το έμαθα αυτό. Θα το παρουσιάσει η Μπενεντέτα Τουρίν το σχέδιο έχει σκοπό να ενθαρρύνει τους νέους που κατάγονται από όλη την Ευρώπη να ε, βοηθήσουν ε, την ένταξη των, ε, και την αφομοίωση όλων των προσφύγων. Βλέπω εδώ μια Ιταλική ταυτότητα. Προτείνεται εργαστήρια, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν εθελοντές, διεθνείς αλλά και τοπικές αρχές και τοπικές κοινότητες. Συγχαρητήρια για αυτή την τόσο ευαίσθητη πρωτοβουλία στην οποία πρέπει να δείξουμε πολύ περισσότερα παραδείγματα αλληλεγγύη στην Ευρώπη, η οποία ορισμένε φορέ ξεχνά αυτό το καθήκον τη αλληλεγγύη. Να παρουσιάσω και του υπολείπου. Το δεύτερο βραβείο είναι το Αναζητώντα τον Καρλομάγνο, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και πολύ ευχάριστο πρέπει να πω από την Ελλάδα. Είναι η χώρα καταγωγής, ε, η Χαρίκλια Μπλουγκούρου, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον διότι είναι ένα σχέδιο ε, ε, μαθητών ενός λυκείου στον ε, πύργο που δημιούργησαν ένα βιντεοπαιχνίδι για τον Καρλομάγνο το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο εντάσσεται στην πολιτιστική κληρονομιά κατά την άποψή μου αναγνωρίζεται ως πατέρας της Ευρώπης γιατί προσπάθησε να δημιουργήσει την Ένωση συγχαρητήρια αν θέλετε μπορείτε να βάλετε ακουστικά και να προσπαθήσετε να δείτε ε, πού βρίσκεται η γλώσσα σας, τι γλώσσα προτιμάτε. Τα Ιταλικά είναι στο 4. Και στο τρίτο βραβείο έχουμε τον Τίλμαν Χάιντελκ Young European Council από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Νέων είναι μια ετήσια ε, διεθνής διάσκεψη που ενώνει ε, νέους ε, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασιζόμαστε βέβαια στους νέους από το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή και ο στόχος είναι να συνεισφέρουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Πρόκειται για μια επιλογή η οποία έγινε από κριτική επιτροπή που διάλεξε τρεις τελείως διαφορετικές προτάσεις αυτή είναι και η ε, αξία αυτού του βραβείου και τρεις πολύ ενδιαφέρουσες χώρες, διότι με τελείως διαφορετικό τρόπο συμμετέχουν σε διαδικασίες και τελείως διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις. Έχουμε περίπου μια ώρα λοιπόν για να παρουσιάσουν τα παιδιά τις ε, προτάσεις τους και να συζητήσουμε. Ο καθένας από εσά έχει 7 λεπτά στη διάθεσή του και από εκεί και πέρα θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους. Δεν έχουν μείνει πολλές ε, ημέρες εργασίας. Έχουμε το απόγευμα ένα πολύ ε, σημαντικό ε, ε, γεγονός, μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Δεν έχουμε πολλούς συναδέλφους εδώ, αλλά θα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Να δώσω αμέσως λοιπόν το λόγο στην Πεντατουρίν από το Integrate. Παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους. Ε, θα μιλήσω για το πρόγραμμα Integrate. Ε, πώς μπορώ να αλλάξω τη διαφάνεια, πείτε μου παρακαλώ. Θα σας παρουσιάσω σύντομα τι κάνουμε εμείς ως ΑΕΖΕΚ. Είμαστε μία μη πολιτική οργάνωση για την αποφυγή των διακρίσεων. Είναι η μεγαλύτερη φοιτητική οργάνωση στον κόσμο και δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να αποφευθούν οι συγκρούσεις όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και μία ομάδα φοιτητών στην Ευρώπη αποφάσισαν ότι ήθελαν να ε, υπάρχει η ειρήνη και ε, η ε, ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ανθρώπων. Θέλησε λοιπόν ένα καλύτερο μέλλον για την νεολαία και γι' αυτό ήθελε να δημιουργήσει νέους ηγέτες και τέσσερα στοιχεία υπάρχουν ε, εδώ που είναι το να εμπνέει κανείς άλλους, ε, το ε, να μπορεί να λάβει ηγετική θέση κλπ. Λοιπόν, με πραγματικές πολιτιστικές αλλαγές θέλησαμε να το πετύχουμε αυτό. Στην Ινδία το 2015 είχαμε το διεθνές, ε, τη διεθνή διάσκεψη της ΆΙΖΑΚ όπου συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι από όλο τον κόσμο. Και οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι συναντήθηκαν για να συνειδητοποιήσουμε τι είδους πρόγραμμα θέλουμε να δημιουργήσουμε που να αντιμετωπίζει ευρωπαϊκά θέματα. Και από τους νέους που συγκεντρώθηκαν εκεί. Ε, είδαμε ότι θέλουμε να επικεντρωθούμε στην ένταξη των ε, άσυλων και μεταναστών στην Ευρώπη στην ε, Ιταλία σε μια διάσκεψη κορυφής τον Οκτώβριο του 2015 με όλους τους εκπροσώπους της Ευρώπης ε, ε, ξεκίνησε το πρόγραμμα. Στόχο λοιπόν έχει να δημιουργεί επαφές μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων, τοπικών κοινοτήτων και ευρωπαϊκών φοιτητών οι φοιτητές ε, πηγαίνουν ε, στους ε, καταβλισμούς των προσφύγων όπου διδάσκουν, βοηθούν, ψυχαγωγούν κλπ. Και το κάνουμε αυτό όχι μόνο για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες και τους ετούντε άσυλο, αλλά θέλουμε και οι Ευρωπαίοι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με την πραγματικότητα και να καταλάβουν ότι είναι, πρόκειται για ανθρώπους από τους οποίους μπορούμε να μάθουμε πράγματα και ότι μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ένταξη των ανθρώπων αυτών. Η αξία του προγράμματος, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο, είναι ότι θέλουμε οι νέοι φοιτητέ να καταλάβουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι, διότι είναι πολύ ωραίο να συζητάει κανείς, ε, να καταλαβαίνουν ποια είναι τα προβλήματα, αλλά ε, τι μπορούμε να κάνουμε για να τα λύσουμε αυτά. Και στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ εύκολο να ταξιδεύει κανείς. Θέλουμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε τους νέους να πάνε σε, άλλους χώρους, σε άλλες χώρες και να βοηθήσουν στην ένταξη ε, προσφύγων και τούντων άσυλο. Τους ε, καλούμε λοιπόν ε, να μην περιμένουν να γίνει η ένταξη από μόνη της. Πηγαίνουμε εμείς επί τόπου και το κάνουμε αυτό. Έβγαλα φωτογραφίες. Βλέπετε εδώ μία νέα από την Ισπανία που πήγε στην Επαβία. Βλέπετε από πίσω κρύβεται μια άλλη φωτογραφία, κάτι μάλλον πήγε στραβά. Ε, συμμετείχαν και άνθρωποι από την Αυστρία. Είχαμε και ένα βίντεο, δεν ξέρω αν λειτουργεί, μια Γαλλίδα διδάσκει Ιταλικά σε πρόσφυγες και είναι πολύ ωραίο αυτό διότι ε, γελάνε, κάνουν αστεία για την Ιταλική γλώσσα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εδώ και ένα χρόνο έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα. Ξεκίνησε όμως από εδώ. Ξεκίνησε στην Ιταλία δηλαδή. Η Ιταλία πρόθεσε το πρόγραμμα αυτό. Δημιουργήσαμε λοιπόν, ε, οργανώσαμε τη διάσκεψη, συνεργαστήκαμε με την Άιζακ και αυτή τη στιγμή πάνω από 10 χώρες στην Ευρώπη συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Συμμετέχουν δηλαδή μη κυβερνητικέ οργανώσει των χωρών αυτών. Οι φοιτητέ όμω που συμμετέχουν προέρχονται από το σύνολο τη Ευρώπη και συχνά και έρχονται και εκτό Ευρώπη. Ε, θέλουν και άλλες χώρες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και Έχουμε λάβει και αιτήματα από τους ε, καταβλισμούς ε, προσφύγων που ζητούν βοήθεια. Για παράδειγμα, είχαν ένα πρόγραμμα στο Μπάρι της Ιταλίας. Γνωρίζετε ότι η Ιταλία ε, επηρεάζεται πολύ περισσότερο από το θέμα αυτό από ότι άλλα μέρη. Παρ' όλα αυτά έχουμε προγράμματα σε πολλά μέρη. Κάθε δύο μήνες έχουμε νέους εθελοντές για τους καταβλισμούς. και όλο και περισσότεροι φορείς που συμμετέχουν στην ΑΙΕΖΕΚ θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό και από την Τουρκία είχαμε θετικά μηνύματα από την νεολαία. Μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε τα πρώτα μετρήσιμα επιτέχματα του προγράμματος αυτού για να δούμε πόσο έχει βοηθήσει τους φοιτητές και τις τοπικές κοινότητες το πρόγραμμα αυτό διότι πέρα από τα εργαστήρια έχουμε και προγράμματα που, όπου συμμετέχει και η τοπική κοινωνία. Ο πρόεδρος ε, της Άιζεκ πήγε στην ε, Αυστρία για ένα πρόγραμμα ένταξης ε, όπου διδάσκανε οι πρόσφυγες τους τους ντόπιου, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό αυτό που βλέπουμε συνήθω. Συνήθω εγώ ως ε, θελόντρια ε, διδάσκω τους πρόσφυγες. Ε, βλέπουμε όμως ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων. Αυτά από μένα. Very, very Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση και νομίζω ότι γνωρίζετε ίσως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την ε, προστασία των ε, παιδιών προσφύγων και για την ε, βοήθεια προς αυτούς, αυξάνεται ο προπολογισμό και ανοίγει και τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικές διόδους, ώστε τα παιδιά πρόσφυγες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και να τα υποστηρίξουμε για να μην έχουμε μια χαμένη γενιά. Υπάρχει λοιπόν κατάλληλη προσοχή ε, σχετίζεται λοιπόν και το θέμα σας με αυτό και το γεγονός ότι είστε εσείς πρωταγωνιστές ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και όμορφο. Να περάσω στο δεύτερο βραβείο, γιατί είναι δεύτερο βέβαια, αλλά πάλι βραβείο είναι, η Χαρίκλια Μπλουγκούρου, αναζητώντας τον Καρλομάγνο. Αυτό το ε, ελληνικό βίντεο παιχνίδι για τον Καρλομάγνο που μας ενδιαφέρει πολύ. Θα μας δείξετε και ένα κομματάκι. Ε, ναι, φυσικά θα σας δείξω ένα κομμάτι. Ε, λοιπόν, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως νέοι που ενδιαφέρονται για την Ενωμένη Ευρώπη και ρομαντίζονται μια Ευρώπη των λαών και των πολιτισμών, δημιουργήσαμε ένα παιχνίδι ρετοαπαντήσεων για την Ευρώπη στα χρόνια του Καρλομάγνου και σήμερα. Ε, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η ιδιαίτερη εκπαίδευση, λόγω της οικονομικής κρίσης και των διαφόρων άλλων προβλημάτων της, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων και να κατακτήσουμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή διάκριση στο βραβείο Καρλομάγνου για την νεότητα 2015-2016. Ε, σε μια λαμπρή... Συγγνώμη. Σε μια λαμπρή τελετή που έγινε στο Άχιν της Γερμανίας, από όπου και κατάγει το Καρλομάγνος, πατέρας της Ευρώπης. Το παιχνίδι που δημιουργήσαμε αποτελείται από μία μακέτα χάρτη, κάρτες και ζάρια. Κάθε κάρτα περιέχει ερωτήσεις και κάθε παίκτη πρέπει να τις απαντήσει. Εάν απαντήσει σωστά, ρίχνει το ζάρι το οποίο του υποδεικνύει σε ποια πόλη να συνεχίσει. Με το χρηματικό έπαθλο αναβαθμίσαμε το παιχνίδι από επιτραπέζιο σε ψηφιακό, με σκοπό όλοι να μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο και να παίξουν την ψηφιακή αυτή εφαρμογή. Στόχος του παιχνιδιού είναι να μάθει στους νέους ότι δεν υπάρχει ήττα. Στο παιχνίδι μας δεν υπάρχει νικητής. Είναι ένα παιχνίδι γνώσεων που στοχεύει στην εκμάθηση νέων πληροφοριών για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ακολουθήσει τον Καρλομάγνο στα πατρικά του εδάφη. Να ζήσει στην καρολίκη εποχή και μαζί του να τον βοηθήσει με τις κατακτήσεις του. Το παιχνίδι περιέχει έξι τυχαίες πόλεις που κατέκτησε ο Καρλομάγνος και σε κάθε πόλη υπάρχει ένα μήνυμα που δίνει πληροφορίες για το συγκεκριμένο μέρος. Στη συνέχεια υπάρχει μία ερώτηση και ο παίκτη, ένα απαντήσει σωστά, παίρνει ένα πόντο. Ανάλογα με τους πόντους που θα συλλέξει, παίρνει έναν τίτλο, ή του υπηκόου, ή του χωρικού, ή τον τίτλο του Καρλομάγνου. Όπως τόνισα και νωρίτερα, το παιχνίδι δεν έχει στόχο τη νίκη, αλλά την γνώση. Ελπίζουμε να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση σε όλα εκείνα τα νέα παιδιά που προσπαθούν να αγωνίζονται καθημερινά για κάτι καλύτερο και να μην παρατούνται από τις προσπάθειές τους, να συνεχίσουν μέχρι το τέλος όσα εμπόδια και αν βρεθούν στο δρόμο τους. Γιατί πάντοτε αυτό το ταξίδι έχει να τους προσφέρει πολλά, όπως λέει και ο ποιητής Καβάθης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δεν θα μας δείξει το παιχνίδι, ε. δεν μπορούμε να το δούμε. Εντάξει για να έχουμε μια ιδέα. Θα σας δώσω αργότερα κάποιες κάρτες. Ωραία, γιατί φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στο τρίτο βραβείο, ο Τίλμαν Χάιντελκ από το Young European Council του, Ευρω... του Ηνωμένου Βασιλείου ε, και θα μας πει περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κώστα για την πρόσκληση και φυσικά για το καλωσόρισμα και για την Οργανωτική Επιτροπή του Βραβείου Καρλεμάρνου. Είναι τιμή που βρισκόμαστε εδώ. Θα αναφερθώ στο τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη διάσκεψη, ε, από πού ξεκινήσαμε, μπορείτε να δείτε και τις διαφάνειες. Μετά θα σας αναφέρω τη διάσκεψη και την ε, εξέλιξη και τι έγινε από τότε που λάβαμε το βραβείο ο οργανισμός ε, πίσω από το Young European Council ε, λέγεται Young European Leadership. είμαστε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που εδρεύει εδώ στις Βρυξέλλες. Ξεκινήσαμε το 2011 ε, διότι πιστεύουμε ότι πρέπει οι νέοι να είναι μια αντιπροσωπευτική ομάδα στην Ευρώπη. Ε, πρέπει να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τις πολιτικές αποφάσεις γιατί δεν επηρεάζονται αυτή τη στιγμή και θέλουμε να τα αλλάξουμε αυτό. Πρέπει να έχουμε μια ισχυρή φωνή οι νέοι για να έχουν τα μέσα και την πρόσβαση να χτίσουν το μέλλον της Ευρώπης. Η ομάδα που βρίσκεται πίσω από το Young European Leadership ε, αποτελείται από 30 εθελοντές από 16 χώρες αυτή τη στιγμή. Αλλάζει βεβαίως διότι είναι ομάδα εθελοντών και επιτυχάνουμε τους στόχους μας επειδή επικεντρωνόμαστε σε δύο πράγματα. Υπάρχει ένα ε, πρόγραμμα παγκόσμιων αντιπροσωπιών. Ε, συμμετέχουμε σε διεθνείς ε, διασκέψεις. Η πιο διάσημη είναι ο εταίρος των νέων του G20. Ε, έχουμε επίσης μια αντίστοιχη ομάδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και προσπαθούμε να μιλήσουμε απευθεία με τον Ομπάμα, τη Μέρκελ και τα άλλα μέλη του G20 και επίσης έχουμε και άλλα προγράμματα, το Young European Council, το οποίο θα σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες. Το Young European Council, ε, η YEC, είναι μια διεθνή διάσκεψη νέων, η οποία ε, διεξάγεται κάθε χρόνο, ώστε να δώσουμε στους νέους τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και νετόεμες αλλά ρεαλιστικές προτάσεις ε, πολιτικής στους πολιτικούς ηθήνοντες. Αυτό γίνεται μέσω άμεσης πρόσβασης σε ηθήνοντες όπως εσείς, ευρωβουλευτές, αλλά και επιτρόπους, πρέσβεις και ε, είναι λίγο απλά τα πράγματα. Καταρχάς υπάρχει μια διαδικασία ε, ε, τήσεων που μπορεί να έχει τη συμμετοχή όλων και επίσης δεχόμαστε φύσεις ιδέες να του, μας πούνε οι άνθρωποι πώς θεωρούν ότι πρέπει να διαμορφωθεί η Ευρώπη. μετά, στη διάσκεψη υπάρχει μια εβδομάδα διαπραγματεύσεων όπου οι νέοι άνθρωποι οργανώνονται σε συμβούλια ε, που επικεντρώνονται σε θέματα όπως ισότητα φύλων, κοινωνική ένταξη, πολιτικές ε, ολοκλήρωσης, ε, η μετάβαση από την παιδεία στην απασχόληση και το καθεξής και ο καθένας εκπροσωπεί τη χώρα του. Δηλαδή εκπρόσωπος από τη Σλοβακία εκπροσωπεί τη Σλοβακία, αλλά όχι την άποψη της κυβέρνησης, αλλά την προσωπική του άποψη, ώστε να έχουμε νέες ιδέες, διότι δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε αυτά τα οποία υπάρχουν ήδη, αλλά χρειαζόμαστε νέα όθηση, νέα οράματα για την πρόθεση της Ευρώπης. Στη διάρκεια της διαδικασίας συνδέουμε τους νέους ανθρώπους με ενδιαφερομένους, για παράδειγμα τους καλούμε για συναντήσεις ε, ε, και μπορούν να συζητήσουν τι ακριβώς υπάρχει, τι ε, σκέφτονται οι νέοι. Υπάρχει επίσης μια διαδικασία ε, προσέγγισης των ενδιαφερομένων. Για παράδειγμα, στην τελετή λήξης φέτος είχαμε προσκαλέσει τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, την Αντιπρόεδρο, την κυρία Γεωργίεβα, και μας ε, μίλησε, συζήτησαν τα παιδιά της ιδέες τους μαζί τους. Δεν είναι πράγματα λοιπόν τα οποία καταλήγουν σε ένα χαρτί το οποίο θα πάει σε ένα σιρτάρι και θα χαθεί. Ε, τα επιτεύγματά μας είναι καταρχάς ότι υπάρχει διάλογος μεταξύ γενεών και μεταξύ διαφόρων τομέων. Δεύτερον, το βραβείο νέων Κάρλο Μάγνος που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για μας γιατί αναγνωρίζετε το εθελοντικό μας έργο και ε, εμείς ε, εργαζόμαστε ανοιχθημερών για το θέμα αυτό ενώ την ημέρα ε, δουλεύουμε ή σπουδάζουμε ούτω καθεξής και φυσικά ε, υπάρχει και η ε, χορηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο ευχαριστούμε. Ε, βεβαίως δεν θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί αυτή η διάσκεψη μεταξύ την υποστήριξη των χορηγών μας, τον Πόντιο, τα ξενοδοχεία Μένιγκερ, τα ξενοδοχεία των, ε, τους ευρωβουλευτές, την Τζούλι Ward, η Μίριαμ Ντάλι και άλλοι που δεν είναι εδώ σήμερα βεβαίω. Τώρα, τι γίνεται με ε, το ευρύτερο πλαίσιο. Καταρχάς το πρόγραμμα είναι πενταετές. Η ιδέα ξεκίνησε το 2013, μάλιστα με κάτι συναδέλφου καθόμασταν σε ένα μπαρ ένα βράδυ και κοιτούσαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώ μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα να επικεντρωθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ανάπτυξη τη Ευρώπη. Αυτή ήταν η πρώτη ιδέα. Το 2014 είχαμε την πρώτη έκδοση του Young European Council. Ε, προσδώσαμε κάποια ουσία, αυξήσαμε τον αριθμό των συμμετεχόντων, των ομιλητών που μπορούσαμε να προσκαλέσουμε και τη γενικότερη προσοχή ε, και προβολή του προγράμματος. Το 2016 και από τότε που λάβαμε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνος, ε, το πρόγραμμα ε, θα διεξαχθεί βεβαίως και φέτη, φέτος και αυξήσαμε λίγο την δομή. Έχει πλέον δομή αντίστοιχη με τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια που γίνονται εδώ στις Βρυξέλλες ή ε, στις χώρες μέλη. Έτσι έχουμε κάτι που είναι ρεαλιστικό αλλά με τελείως διαφορετική συνεισφορά. Έχουμε αυξήσει την προσέγγιση των ενδιαφερομένων. Θα πρέπει πλέον οι άνθρωποι να γνωρίζουν τις ιδέες των νέων ανθρώπων και έχουμε αυξήσει τον αριθμό των ετούντων, των συμμετεχών δηλαδή έχει ε, γίνει γνωστό το πρόγραμμα. Είναι βέβαια ένα πρώτο βήμα της διαδικασίας, το 2017-2018 θα ε, επικεντρωθούμε στην πρόσβαση στο πρόγραμμα, ώστε όποιος θέλει να κάνει αίτηση, όποιος θέλει να συμμετέχει, να μπορεί να συμμετέχει και να μην ε, έχει σχέση με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, αλλά με τη διάθεση να συμμετέχει. Επίσης ε, ε, έχουμε ένα πρόγραμμα με την ε, Προεδρία του Συμβουλίου. Φέτος συνεργαζόμαστε με το Τρίο των Προεδιών. Είχαμε εκπροσώπους από την Ολλανδία και τη Μάλκτα και τη μελλοντική Προεδρία της Εστονίας. Είχαμε τους πρέσβεις παρόντες εκεί, ώστε να μπορέσουμε να συντονίσουμε το πρόγραμμά μας με το πρόγραμμά τους. Επίσης είμαστε πεπισμένοι ότι οι νέοι είναι ο μοχλός της αλλαγής στην κοινωνία μας. Είναι οι άνθρωποι που θα είναι εδώ αύριο, αλλά είναι και το σήμερα. Επομένως πρέπει να συμμετέχουμε έχουν οι νέοι, είναι η ρίζα της κοινωνίας μας και γι' αυτό ακριβώ θέλουμε να έχουμε μεγάλη συμμετοχή της κοινωνίας ώστε να ακούγεται η φωνή όλων. Και τώρα θα ήθελα να ολοκληρώσω με μια πρόσκληση. Το ε, πρόγραμμά μας θα γίνει και φέτος το Νοέμβριο με την ε, βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα έχουμε την κυρία Γεωργίεβα, την κυρία Μπονίτσι και τον κύριο Ντεγκόιερ. Αν θέλετε να έρθετε θα υπάρχει ένα γεύμα ε, που θα μπορέσετε να ε, συναντήσετε και τους ε, καλεσμένους μας. Αν ενδιαφέρεστε μπορώ να σας δώσω όλες τις πληροφορίες και με χαρά θα σας υποδεχθούμε σε αυτό το γεύμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή διότι ε, περιλαμβάνει τόσους πολλούς νέους αλλά και ε, για τον ε, ε, διάλογο μεταξύ γενεών που προτείνει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Τρία εξαιρετικά προγράμματα πρέπει να πω, τα οποία άξιζαν να κερδίσουν και ίσως ε, θα μπορούσαν να προβληθούν και λίγο περισσότερο. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν και μια προθήκη στην οποία θα παρουσιάζουμε τα έργα μας, να είναι υπόδειγμα ε, το οποίο θα μπορούσε να ε, ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν παρατηρήσεις από πλευρά συναδέλφων ή η κυρια Φερχάιερ. Καταρχάς, θα ήθελα να σας, να σας ευχαριστήσω για την αφοσίωσή σας. Χρειαζόμαστε νέους που μπορούν να προωθήσουν την Ευρώπη, που μπορούν να ασχοληθούν με την Ευρώπη. Χαίρομαι ιδιαίτερα επειδή είμαι από το Άχεν, είμαι βουλευτής του Άχεν. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς αλλά και όλους τους άλλους που ε, συμμετείχαν στον διαγωνισμό αυτόν, αλλά ε, και πολλούς νέους που ε, παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες σε όλη την Ευρώπη που δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Συχνά δεν ε, αρκούν και οι πόροι για να χρηματοδοτηθούν όλες αυτές ε, οι πρωτοβουλίες, αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ πόσο σημαντική είναι η δουλειά που κάνετε, πόσο σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες των νέων, ώστε να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους ανθρώπους, πιο κοντά στους νέου. Χωρίς τη δική σας συμμετοχή δεν θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα μέλλον για την Ευρώπη. Και είναι πολύ σαφής η πολυμορφία των ε, πρωτοβουλειών, ε, βλέποντας ε, και μόνο τους βραβευμένους, διότι έχουμε το ένα πρόγραμμα για την ένταξη, έχουμε ένα πρόγραμμα για την ευρωπαϊκή ιστορία και είναι πολύ σημαντικές οι πτυχές αυτές για την Ευρώπη. Θέλουμε να φέρουμε τους νέους σε επαφή με την Ευρώπη, διότι πολλά από αυτά που έχει πετύχει η Ευρώπη δεν είναι η ιστορία, είναι και η καθημερινή μας ζωή. Λειτουργούν όλα, μπορούμε να τα ταξιδέψουμε, δεν το προσέχουμε, δεν το εννοώ αυτό ε, αρνητικά, αλλά ιδιαίτερα γι' αυτό μου αρέσει ε, η πρωτοβουλία που ε, έχει να κάνει με την ιστορία. Πώς φτάσαμε εδώ και Είδαμε τόσους πολέμους στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των αιώνων. Ενώ σήμερα λύνουμε τα προβλήματά μας με τη συζήτηση με ε, πολιτικούς ε, δημοκρατικούς θεσμούς. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τα διατηρήσουμε αυτά και χρειαζόμαστε νέους όπως ε, εσείς για να καταπολεμήσουμε και τις ακροδεξιές τάσεις που βλέπουμε στους, ε, σε μερικούς νέους. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για τις προσπάθειές σας. Ευχαριστώ την Σαμπίνε. Η κυρία Κάμερεβερτ. Ja, vielen herzlichen Dank, Silvia. Ευχαριστώ πολύ, Σίλβια. Μπορώ να συμφωνήσω μόνο με την συνάδελφό μου την Σαμπίνε Φερχάγενε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω ε, θερμά για τις προσπάθειές σας. και που προσπαθείτε να ε, διατηρήσετε στη ζωή και να αναπτύξετε περαιτέρω τις πρωτοβουλίες ε, τις οποίες ξεκινήσατε. Η Ευρώπη χρειάζεται τέτοιες πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους. Κατά την ε, τελευταία απονομή του βραβείου Κάρλε Μάγνου είπα στους ε, Γερμανούς εκπροσώπους ότι είναι τόσο ε, ενδιαφέροντα όλα τα προγράμματα, θα έπρεπε να ε, βραβεύσουμε όλες τις πρωτοβουλίες. Ουσιαστικά εκπροσωπείτε τους τόσους νέους στην Ευρώπη που αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Και όταν βλέπω τέτοια προγράμματα δεν ανησυχώ για το μέλλον της Ευρώπης. Παρότι αυτή τη στιγμή Μερικέ φορές μπορεί να έχει κανείς αρνητική αίσθηση όσον αφορά τις εθνικιστικές τάσει που, ε, που βλέπουμε παντού στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αν ακόμα περισσότεροι νέοι ε, ασχοληθούν με πρωτοβουλίε όπω τι δικέ σα, δεν θα πρέπει να ανησυχούμε για το μέλλον τη Ευρώπη. Οι πρωτοβουλίε σα είναι πολύ διαφορετικέ μεταξύ του ε, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η πρωτοβουλία ε, που συνδέεται με την ιστορία, διότι νομίζω ότι μπορεί κανεί να οικοδομήσει το μέλλον μόνο αν γνωρίζει την ιστορία του και συνειδητοποιήσει τα λάθη που έχουν γίνει στην ιστορία για να αποφύγει στο μέλλον να γίνουν τα ίδια λάθη και να μπορέσουμε μαζί να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Και εμένα μου άρεσε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, ε, αυτή η πρωτοβουλία σας, αλλά όλες ε, μου άρεσαν και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω με εξίσου πολύ αφοσίωση να συνεχίσετε ενδεχομένως ε, να δημιουργήσετε νέα προγράμματα, νέες πρωτοβουλίες και στο όνομα της πολιτικής μου ομάδας θα ήθελα να σας ευχηθώ ότι καλύτερο για το μέλλον. Συνεχίστε τις προσπάθειές σας. Ευχαριστώ. Η Χέλγα Τρίπελ, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τις ευχαριστίες και τους επένους ε, που σας δόθηκαν. Είναι μεγάλη χαρά να έχουμε εδώ σήμερα τους ε, νέους νικητές ε, του βραβείου Καρλομάγνου. Και πέρσι είδαμε εξίσου πολύ αφοσίωση και πάθος ε, για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και οι συνάδελφοι και εγώ χαίρομαι όταν βλέπω νέους που έχουν τη δύναμη, τη διάθεση και το πάθος να ασχοληθούν με τέτοια πράγματα διότι έτσι μπορείτε να ε, καλέσετε και άλλους νέους να συμμετάσχουν και ε, ειδικά σε εποχές όπως είναι η σημερινή που βλέπουμε ότι ε, πολλοί γυρνούν την πλάτη στις κοινέ προσπάθειες Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα, πώς μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε άλλους νέους να συμμετάσχουν, ε, να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να συμβάλλουν ε, θετικά στην ε, καλή εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από μένα λοιπόν σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία στη συνέχεια. Και κάντε ό,τι μπορείτε ώστε όσο γίνεται περισσότεροι να μάθουν τις πρωτοβουλίες σας. Εύχομαι λοιπόν και για σας προσωπικά και για, τα, και για τις πρωτοβουλίες σας ε, κάθε επιτυχία. <clears throat> Ευχαριστώ, Λουίτζι Μόργανο. Και εγώ θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω ε, για τα τρία αυτά προγράμματα, διότι είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντο. Δεύτερον, ε, νομίζω ότι μεταξύ άλλων μας ε, μιλούν για αυτή την περισσότερη εμπιστοσύνη που πρέπει και εμείς ε, να έχουμε στο μέλλον, διότι αποδεικνύουν ότι κάποιες πρωτοβουλίες μας βοηθούν να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και δεσμεύεστε ε, να κάνετε πράγματα. Και το λέω αυτό διότι πολύ συχνά αυτοί που δεσμεύονται σοβαρά για να ε, δημιουργήσουν πράγματα δεν είναι στις ειδήσει. Ε, και αυτό δεν είναι αποτυχία όχι μόνο της επικοινωνίας αλλά και του πολιτισμού μας, τον οποίο πρέπει να ξαναβρούμε. Και νομίζω γιατί ε, μπορέσετε να συμμετέχετε και σε ένα τμήμα της συζήτησης που αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς που θα έχουμε το 2018 ότι το γεγονός ότι κάποιες επιλογές ε, που προκύπτουν από βούληση σαν αυτή που επιδεικνύετε εσείς προκύπτουν από ε, πρωτοβουλίες σαν αυτά τα τρία βραβεία Καρλομάγνου τα οποία γεννιούνται και στη συνέχεια προχωρούν παρά το γεγονός ότι δεν αντιλαμβανόμαστε από την ε, αρχή δημιουργούνται κατάλληλες προϋποθέσεις για να προοδεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε κάτι. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο συνάδελφο που να θέλει το λόγο. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, να πείτε κάτι. ποιο θέλει το λόγο. Να ξεκινήσουμε από τον τελευταίο. Παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπαν οι κυρίες Φερχάιεν, ε, Κάμερα και ε, Τρούιπελ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας, αλλά πράγματι η γνώση της ιστορίας ε, είναι απαραίτητη. Η δική μου, φαμίλ, η δική μου οικογένεια προέρχεται από την ε, Ανατολική Γερμανία. Ε, ζούσαμε πίσω από το τείχος και είμαι ο πρώτος της οι οικογένειές μου που ε, μπόρεσα να φύγω από τη χώρα μου, να φύγω από την ε, Γερμανία, να δω την Ευρώπη. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε τις δυνατότητες αυτές. Ε, αν κοιτάξουμε ακόμα πιο πίσω στην ιστορία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Καρλομάγνο για κάτι θετικό και συμφωνώ με τα όσα είπατε και σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και φυσικά θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τον καλό αυτόν σκοπό. Ευχαριστώ. Ωραία. Η ελπίδα μας είναι το πρόγραμμά σας να συνεχιστεί. Ο Καρλομάγνος ήταν το κίνητρο, αλλά νομίζω ότι εσείς θα συνεχίσετε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κι εσείς κάτι, παρακαλώ. Ε, θέλω να πω ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τα καλά σας λόγια και τις ευχαριστίες σας. Και θέλω να πω ότι δημιουργήσαμε αυτό το παιχνίδι για αυτό το σκοπό. Δηλαδή κάθε παίκτη, κάθε παιδί, κάθε πολίτης να μάθει ε, για τον Καρλομάγνο, για την Ευρώπη και για την ιστορία της Ευρώπης. Θέλουμε μέσα από αυτό το παιχνίδι ε, να γνωρίζουν όλοι για την Ευρώπη και όπως είπα και πριν δεν υπάρχει νικητή σε αυτό το παιχνίδι αλλά στόχος μας είναι η γνώση. Ευχαριστώ και πάλι. Ε, είναι πολύ ωραίο να έχει ένα παιχνίδι ε, στο οποίο ε, αποκομίζει κανείς γνώσεις ε, και αυτή είναι η νίκη κάθε φορά. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στο 2018 που θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, άειλης και ηλικής, αλλά και οποιαδήποτε νέα μορφή λοιπόν μπορείτε να επινοήσετε εσείς και ο κύριος Μόργανο έκανε έκκληση στους νέους για να έχουμε κάτι αντίστοιχο για την πολιτιστική κληρονομιά. Θα μπορούσε να είναι μια ιδέα. Εσεί είστε ένα βήμα μπροστά σε σχέση με του υπόλοιπους. Ε, η κυρία Τουρίν, παρακαλώ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω βεβαίως για τα όσα μας είπατε. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι για μένα το βραβείο Καρλομάχνου είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι ε, δημιουργεί πρότυπα, παρουσιάζει πρότυπα ε, για σωστή ευρωπαϊκή ηθαγένεια ε, που είναι διαφορετικό από την ηθαγένεια που έχει ο καθένας από τη χώρα του. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και φαίνεται από τα προγράμματα. Πώς οι νέοι όλης της Ευρώπης μπορούν να δουν αυτά τα προγράμματα, μπορούν να δουν τι σημαίνει να είναι κανείς ενεργός πολίτης και να έχει ένα πρότυπο σωστής ηθαγένειας που για μένα είναι το πιο σημαντικό. Αυτό το οποίο ονειρεύομαι για την Ευρώπη και για κάθε χώρα στον κόσμο στην πραγματικότητα είναι όλοι, όλη η κοινωνία των πολιτών να έχουν μια ισχυρή αίσθηση ηθαγένειας και να ξέρουν τι σημαίνει να είναι καλός πολίτης. Ε, και αυτό βλέπουμε σε όλα τα προγράμματα του Καρλομάγνου. Ε, ένα πρότυπο για να δουν όλοι τι σημαίνει να είναι καλός πολίτης και να δουν πώς μπορούν από εκεί και πέρα στη συνέχεια να συνεισφέρουν ώστε η Ευρώπη να γίνει μια καλύτερη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια αλλά και για την πρωτοβουλία του Καρλομάγνου που είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για μένα εδώ σήμερα. Ωραία. Νομίζω σήμερα είδαμε την καλύτερη όψη της Ευρώπης αυτή για την οποία εργαζόμαστε. Επομένως, έχουμε κάποια αισιοδοξία, διότι είμαστε μαζί σας, ε, σύμμαχοί σας και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε και ε, προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ιδιαίτερα ισχυρές. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες, εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία και αυτή είναι η δημοκρατική εκπροσώπηση των Ευρωπαίων πολιτών. Προσπαθούμε λοιπόν να σας εκπροσωπούμε όσο καλύτερα. Επομένως, οι δικές σας ιδέες, οι δικές σας προτάσεις είναι κάτι το οποίο δεχόμαστε. Χαιρόμαστε που σας φιλοξενήσαμε εδώ σήμερα και χαιρόμαστε που σας είχαμε εδώ μαζί μας. Ε, ευχαριστώ. Με αυτό ολοκληρώνονται οι εργασίες για σήμερα το πρωί και θα συνεχίσουμε σε πέντε λεπτάκια.